σημερισία διάταξη. Ε, δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή, είπα τη Εκπροσώπηση Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια, για τι εκτοπίσει πληθυσμών και κατεδαφίσει κτηρίων στη δυτική όφη συμπεριλαμβανομένων και έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Η κυρία Μογκερίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ε, συνεχίζει να ασχολείται κατά προτεραιότητα με το ζήτημα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο οι στρατηγικές αυτές συζητήσεις γίνονται πάντα στη βραδινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Ελπίζω να μην στέλνουμε κατά αυτόν τον τρόπο κάποιο πολιτικό μήνυμα. Ξέρουμε ότι η έλλειψη πρόοδου προς την ειρήνη ιδίω στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, οδηγεί σε νέα κλιμάκωση της έντασης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να επιμείνουμε σε μια λύση δύο κρατών. Ακόμα και αν οι Παλαιστίνοι και το Ισραήλ δεν απασχολούν τα πρωτοσέλιδα, θα πρέπει εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολούμεθα συνεχώς με το στόχο αυτόν. Γιατί ξέρουμε ότι η βιωσιμότητα μια λύσης δύο κρατών σε καθημερινή βάση τίθεται να αμφιβόλο. Επομένως είναι σημαντικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτικό μας καθήκον να διατηρήσουμε πάντα εν ζωή τη λύση αυτή. Η επέκταση τώρα των επικισμών θέτουν αμφιβόλο τη λύση αυτή των δύο κρατών, καθώς επίσης και οι κατεδαφίσεις και οι δημεύσει κατοικιών που έχουμε στην Παλαιστινιακή πλευρά, καθώ επίση και η καταστροφή έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να μα απασχολήσει κατά τον ίδιο τρόπο και η επιδείνωση τη διαβίωση των Παλαιστινίων στη δώρα τη Γάζα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι επικισμοί από του Ισραηλινού δεν είναι η μόνη πρόκληση για τη λύση των δύο κρατών. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ προκλήσει, οι οποίε λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις, έχουμε ρητορική μίσους, και κατά αυτόν τον τρόπο δεν καταφέρνουν οι άνθρωποι να διαβιώσουν ειρηνικά. Επίσης η ίδια η ενότητα του Παλαιστινιακού κράτους αυτή τη στιγμή δεν βοηθάω καμία προοπτική ειρήνευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε τους λαούς και από τις δύο πλευρές. Ας έχουμε κατά νου λοιπόν μια σφαιρικότερη εικόνα των πραγμάτων, μολονότι επικεντρωνόμαστε όπως και σήμερα το βράδυ σε ζητήματα πιο συγκεκριμένα. Στο ζήτημα το οποίο εσείς επιλέξετε σήμερα το βράδυ ασχολούμεθα με μια συγκεκριμένη πτυχή Τη της γενικότερης αυτής εικόνας που για πάρα πολλούς λόγους όπως σας είπα δεν είναι ενθαρρυντική αυτή τη στιγμή. Και παρόλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες σε καθημερινή βάση προκειμένου να δημιουργηθεί μια λύση δύο κρατών αποφασίστε σήμερα να, συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα των εκτοπίσεων πληθυσμών και των κατεδαφίσεων κτηρίων. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι το Ισραήλ με τη δράση του προωθεί περισσότερους επικισμούς και όπως ξέρετε οι επικισμοί αυτοί στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αλλά και στα πλαίσια του νοσιακού δικαίου θεωρούνται παράνομοι και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το έχει πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε κατά της πολιτικής επικισμών του Ισραήλ. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν νέοι επικισμοί πέρα από τη γραμμή που προβλέπεται στην Συμφωνία του 1967 και βέβαια έχουμε στραφεί κατά οποιασδήποτε μορφής κατεδαφίσεων αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών ή συγκεκριμένων μειονοτήτων και προφανώς στρεφόμαστε κατά οποιασδήποτε έκφρασης βίας και από τις δύο πλευρές. Και όχι επειδή ενδιαφερόμαστε μόνο για την τήρηση του διεθνούς δικαίου, προφανώς αυτό μας αφορά μεσότατα αλλά και επειδή όλες αυτές οι δράσεις μειώνουν τη δυνατότητα των Παλαιστινίων να χρησιμοποιήσουν τη γη τη δικιά τους, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να γνωρίσουν μια κάποια οικονομική ανάπτυξη και δυνατότητα βιωσιμότητας οικονομικής στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να διευκολύνουμε την οικονομική και κοινωνική ευημερία των, των Παλαιστινίων. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι το δυνατό προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκές ανθρωπιστικέ συνθήκες στην Παλαιστίνη. Εξαιτία όμω των χωροταξικών αυτών πολιτικών του Ισραήλ, κάποιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές θεωρούνται παράνομες σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκαιο και για αυτό το λόγο κατεδαφίζονται οι υποδομές αυτές ή απειλούνται με κατεδάφιση από το Ισραήλ. Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα τηρεί τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση να βοηθούμε τους πιο ευάλωτους οπουδήποτε αυτό απαιτείται. Κάθε φορά λοιπόν που συγκεκριμένα ανθρωπιστικά σχέδια πρέπει να λάβουν χώρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να ζητήσουμε πρώτερη αδειοδότηση από τις αρχές του Ισραήλ. Είναι ανθρωπιστικό μας καθήκον, πολιτικό μας καθήκον να προχωρήσουμε με την ανθρωπιστική αυτή δράση. 5.000 περίπου σπίτια έχουν ε, κατεδαφιστεί, 650.000 άτομα έχουν ε, εκτοπιστεί και ένα μεγάλο ποσοστό των κατασκευών αυτών προέρχονται μάλλον είχαν λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι έχει ξεκινήσει ένας διάλογος διαβούλευσης με το Ισραήλ προκειμένου να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και τα εμπόδια που υπάρχουν στη λύση των δύο κρατών και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τους Παλαιστινίους ιδίω όσον αφορά το ζήτημα των επικισμών οι οποίοι στρέφονται εναντίον του. Χρησιμοποίησαμε τον περασμένο μήνα τον διάλογο αυτό και αυτό το σύστημα διαβούλευση για να μιλήσουμε για το ζήτημα των εκτοπίσεων και των κατεδαφίσεων. Και αυτό φαίνεται επίση και συμπεράσμα του Συμβουλίου που εγκρίναμε τον Ιανουάριο. Μέχρι στιγμή έχουμε λίγα απτά αποτελέσματα. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να συνεχίσουν τον διάλογο για έξι ακόμα μήνες, ζητώντας να υπάρχει ένα άμεσο μορατόριουμ όσον αφορά τις αρνητικές αυτές δράσεις στον τομέα Γ, ιδίως όσον αφορά τις ε, ε, κατεδαφίσεις και τις δημεύσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει για τα ζητήματα αυτά να έχουμε ακόμα και μία κάποια αποζημίωση κάθε φορά που έχουμε κατεδάφιση ή δίμευση κτηρίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι αυτές οι δράσεις ζημιώνουν πάρα πολύ οικονομικά και την όλη περιοχή και βέβαια και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε όμω μόνο για οικονομικέ επιπτώσει. Το πιο σημαντικό είναι το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων αυτών και τι θα γίνει τελικά με το ζήτημα των επικισμών. Ξέρετε ότι μόνο μία ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να μας βγάλει από, την τον αρνητικό αυτό φαύλο κύκλο. Θα πρέπει προφανώς επιτόπου να βελτιώσουμε την κατάσταση, και παράλληλα θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον απότερό μας στόχο. Ολοκληρώνοντας λέω ότι θα πρέπει να δούμε τη σφαιρικότερη εικόνα. Σήμερα επικεντρωνόμαστε σε μια συγκεκριμένη πτυχή η οποία είναι πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική αλλά θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε παράλληλα και στη γενικότερη πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Συνήθως εσείς με το ζητάτε αυτό, σήμερα το ζητάω εγώ από εσά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε καθημερινή βάση για να δημιουργήσουμε μια λύση με δύο κράτη που θα συνεπάρχουν ειρηνικά, σε συνθήκες ασφάλειας, προκειμένου να σταματήσει η διένεξη σε κάθε μέτωπο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με την βοήθεια της Ρωσίας, των ΗΠΑ και των εθνών να καταλήξουμε σε μια έκθεση του κουαρτέτου που θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και που θα περιέχει συγκεκριμένε συστάσει για το πώ θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μπορώ στο μέλλον τις επόμενε εβδομάδε, σε μια επόμενη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συζητήσω μαζί σα την έκθεση αυτή. Γιατί αυτό που το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ προοπτικέ να δημιουργηθούν τα δύο αυτά κράτη, να συνεπάρξουν ειρηνικά στο άμεσο μέλλον. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται σήμερα ονειροπολισία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει το όνειρο αυτό να παραμείνει ζωντανό και θα πρέπει μια μέρα να γίνει πραγματικότητα. Ω Ευρωπαίοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εξέλθουμε από αυτόν τον κύκλο βία που βλέπουμε στην περιοχή. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε πάντα στο στόχο αυτό. Ξέρω ότι μπορώ να στηρίζομαι στη δική σας την υποστήριξη προκειμένου να πετύχουμε το στόχο αυτό και βέβαια θα μπορούμε παράλληλα να επιλύουμε κάθε φορά να συζητάμε επιμέρους πτυχές του ζητήματος. Θα ήθελα να σας ζητήσω σε μια επόμενη σύνοδο της Ολεμίας, Ολομελίας με συγχωρείτε, να συζητήσουμε σφαιρικά το ζήτημα του Παλαιστινιακού μέσω της έκθεσης του κουαρτέτου και να αναφερθούμε και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως η γαλλική πρωτοβουλία να έχουμε μια παγκόσμια σύνοδο και να δούμε κατά αυτόν τον τρόπο πώς μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλουμε προκειμένου να επιληθεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και προκειμένου τελικά να γίνει πραγματικότερη ερνευτική διαδικασία για να οδηγηθούμε σε αυτή τη λύση των δύο κρατών. Ξέρω πολύ καλά ότι όλοι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, όλοι προασπίζουμε τον ίδιο στόχο, αλλά δεν θα πρέπει ο στόχος αυτός να αποτελεί απλό σλόγγαν, θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, σε καθημερινές πράξεις που θα δυναμώνει το στόχο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μογκερίνη. Ξεκινά τώρα η συζήτηση. Ο κύριος Πρέντα πρώτος, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπατή Εκπρόσωπε. Παρουσιάσατε το πρόβλημα που συζητάμε απόψε, το ζήτημα των καταδεφίσεων στη Λωρίδα της Γάζας και το ζήτημα είναι περίπλοκο. Μετά τις συμφωνίες του Όσλο, στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τομέας C, ο τομέας Γ παραμένει υπό τον ε, στρατιωτικό έλεγχο ε, του Ισραήλ και γνωρίζουμε ότι το εκμεταλλεύεται το Ισραήλ για τη δημιουργία παράνομα κατασκευών. Και όπως γνωρίζετε επίσης το Ισραήλ έχει κατηγορήσει πολλές φορές την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρηματοδοτεί την ε, δημιουργία κατασκευών στην περιοχή εκείνη κατά παράβαση των συμφωνιών του Όσλο. Πρέπει λοιπόν όμως να βρούμε μια και έναν κοινό τόπο γιατί όπως αντελήφθη από την παρέμβασή σας, ε, το Συμβούλιο ε, σκέφτεται να δημιουργήσει ε, μια στρατηγική για το ζήτημα των κατεδαφίσεων και να ζητήσει την απροζημίωση μετά από τέτοιες κατεδαφίσεις να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός. Υπάρχει συντονισμό μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων κρατών μελών και θα έπρεπε να βασιστούμε σε αυτόν και να τον αναπτύξουμε. Βεβαίω το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσει η ερευνευτική διαδικασία, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται εμπιστοσύνη και από τι δύο πλευρέ. Του τελευταίου μήνε, η πλευρά των Ισραηλινών ε, έχει την αίσθηση ότι τονίζουμε την έλλειψη εμπιστοσύνης, ότι τους δίνουμε το μήνυμα ότι δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα στην περιοχή. Ξέρω ότι αυτά που λέω θα δυσαρεστήσουν τους φίλους μας από την άκρα αριστερά, χωρίς να θέλουν να υπονοήσουν ότι υποστηρίζουν τους τρομοκράτες, αλλά παρόλο αυτά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα στην περιοχή. Θα σε ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε Πρόεδρε. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος Μποστινάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ δεν είναι καινούρια πράγματα τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τα όσα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη οι καταστροφές αυτές από πλευρά των Ισραηλινών πρέπει να καταγγελθούν γιατί κάθε καταστροφή καταστρέφει τη, τους λίθους με τους οποίους θα χτιστεί, θα δημιουργηθεί ο οίκος της ειρήνης, η, η ειρήνη ίδια. Δεν πρόκειται μόνο για τη διάσωση ε, χρημάτων φορολογουμένων της Ευρώπης που έχουν διατεθεί για αυτά τα κτίρια τα οποία καταστράφηκαν. Πρόκειται όμως για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Παλαιστινίων. Αυτά λοιπόν πρέπει να καταλήγουν τα χρήματα αυτά σε εκείνους που πρέπει να υποφεληθούν από αυτά και στους οποίους ανήκουν. Φυσικά είναι προτεραιότητα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής να προαχθεί η ειρηνευτική διαδικασία και να επανεγγραφεί στην ημερήσια διάταξη όπως αναφέρθηκε και από την ύπατη εκπρόσωπο. Πρέπει η βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί ώστε έτσι να καταλήξουμε στη διευθέτηση της μεγαλύτερης σε διάρκεια ιστορικά κρίσης και αντιπαράθεσης ε, ώστε να υπάρξει ειρήνη. Έχουμε υποχρέωση ώστε στον ανθρωπιστικό τομέα να τηρηθούν αυτές οι αρχές. Το Ισραήλ είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους μας. Μία από τις λίγες χώρες με τις οποίες έχουμε μια ολοκληρωμένη και πολύ καλή συνεργασία. Όμως ε, θα πρέπει πέρα από τα δικαιώματά του και τις ασυλίες του το Ισραήλ να αναγνωρίσει ότι έχει καθήκοντα και υποχρεώσεις να τηρεί τα, τις διεθνείς συμφωνίες και τις αρχές ε, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράξει πολλά σε αυτή την περιοχή του κόσμου και θετικά. Σήμερα είναι τόσο σημαντικότερο να συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος να υπάρξει αυτή η επένδυση. Στη συνέχεια για δύο λεπτά ο συνάδελφος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. με την τα όσα συμβαίνουν στον τομέα γάμα με τις, ε, ε, με, με την, ε, τις επεκτάσεις κτηρίων παραβιάζεται η κατάσταση δικαιωμάτων και εδώ υπό την απόκρυψη των πράξεων υπό την ανθρωπιστική βοήθεια παραβιάζονται αυτές οι αρχές. Αυτή η μονομερής δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περιοχή του κόσμου αναζωπυρώνει την κρίση και εδώ φυσικά γίνεται και κατάχρηση κονδυλίων των ε, φορολογουμένων της Ευρώπης. Γι' αυτό κατεπηγόντως πρέπει να ζητήσουμε να τερματιστεί οποιαδήποτε υποστήριξη και χρηματική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, δημιουργία κτηρίων και επεκτάσεων αυτών. Κυρία Μογκερίνη, σε μια χρονική στιγμή όπου από την φόρο τιμήσε το Ισραήλ στα εκατομμύρια θύματα που είχε ε, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου πολέμου πολέμου δεν μπορεί να υιοθετεί μια τέτοια στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζεται η Χαμάς ε, και να γίνεται λόγος για δύο κράτη. Δεν άκουσα ε, να γίνεται λόγος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρόλο της Χαμάς. Αυτό είναι ανεύθυνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεθεί στο περιθώριο και δεν μπορεί να ε, προωθήσει ένα δίκαιο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπέλλερ. Στη συνέχεια Βότμανς παρακαλώ. Η κυρία Βότμανς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε. Από πλευράς μου πρέπει να πω ότι εσείς καταστήσατε σαφές ότι κάνουμε λόγο για την καταστροφή κτηρίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα, αλλά ας παραμείνουμε σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύμμαχος του Ισραήλ και το γνωρίζουμε αυτό. Εν τω μεταξύ εδώ κάνουμε λόγο για να τερματιστούν καταστροφές. Ποτέ δεν είδαμε τέτοια μεγάλη κλίμακα καταστροφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, 75 κτίρια καταστράφηκαν που χρηματοδοτήθηκαν χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Και αυτό είναι ένα κλάσμα μόνο των καταστραφέντων κτηρίων με σύνεση πρέπει να αναφέρεται αυτό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει συστηματική πολιτική διακρίσεων εις βάρος των Παλαιστινίων. Και όλα αυτά φυσικά υπονομεύουν την ιδέα δύο κρατών σε αυτή την περιοχή του κόσμου, πράγμα το οποίο αναφέρατε. Κυρίες και κύριοι, σχολεία, παιδικές χαρές, ήλια ε, πάνελ. Όλα αυτά καταστρέφονται. Αυτά είναι απαράδεκτα. Έχουν χρηματοδοτηθεί από το Βέλγιο, την Ολλανδία. Όλες οι χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν την, τους Παλαιστίνιους. Όμως καταστρέφονται όλα αυτά τα δημιουργία, δημιουργήματα από τους αλαζόνες ε, στρατοκράτες στρατιωτικούς του Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι εκτοπίζονται άνθρωποι. Γνωρίζουμε ότι 400 παιδιά είναι άστεγα σαν αποτέλεσμα αυτών των καταστροφών. Παρόλα αυτά όμως τηρούμε συγγύνη χθείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι απαράδεκτο. Κυρία Μογκερίνη, η Ευρώπη πρέπει να εμείνει και να επιμείνει το ανθρωπιστικό δίκαιο να είναι σεβαστό. Αμφότεροι και οι δύο το τονίζω, Ισραηλινοί και Παλαιστινοί πρέπει να σέβονται τις αρχές του ανθρωπιστικού ε, δικαίου. Θα ήμουν ευγνώμονας αν θα μπορούσατε να μας δώσετε στοιχεία πόσα από αυτά τα κτίρια χρηματοδοτήθηκαν από εμάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία αυτής της χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε κυρία Βάρτμαν. Για 1,5 λεπτό η κυρία Άντερσον παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη μπορεί μέχρι και να μυρίσει κανείς την οσμία από τη σκόνη αυτών των κτίριων όταν έχουμε κατεδαφίσεις πάνω από 500 ε, σπιτιών ε, Παλαιστινίων και αυτές μόνο κατά τη διάρκεια του 2015. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν εμπόδιο στην εξέφρεση μιας ειρηνευτική ε, ειρηνή ε, ε, στην περιοχή. Είναι μέρος μιας στρατηγικής του Ισραήλ η οποία θέλει να διευκολύνει του παράνομου επικισμού. ξεκίνησε το 2015 ο λεγόμενος δομημένος διάλογος, ο οποίος θα είχε μια προθεσμία έξι ε, μηνών και μετά από ε, ένα μήνα δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο την διαπίστωση ότι το Ισραήλ περιφρονεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εντείνει μάλιστα τις ε, επιχειρήσεις καταδαφίσεων. Με, καταστρέφοντας σχολεία με βουλντόζες, καταστρέφοντας υδραγωγία, καταστρέφοντας αποθήκες τροφίμων Μπορούμε να ακούσουμε τους Παλαιστίνιους και την κραυγή αγωνίας τους. Αλλά δεν έχει νόημα για αυτούς γιατί ξέρουν ότι η απάντηση δεν θα βρεθεί ούτε τώρα ούτε σε έξι μήνες. Πρέπει να σταματήσει πλέον η ατιμορρησία του Ισραήλ και πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζονται οι Παλαιστίνοι είναι τη βοήθειά μας, χρειάζονται πράξεις και όχι λόγια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντερσον. Για 1,5 λεπτό η κυρία Άουκεν παρακαλώ. Ναι, Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ισραήλ όντως έχει κατεδαφίσει κτίρια, έχει κατεδαφίσει δεξαμενές, έχει κατεδαφίσει σχολεία, σχολικές τάξεις, υδροελεκτρικά κέντρα. Πάνω σε όλα αυτά τα κτίρια πολλές φορές σχηματίζει ακόμα και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολλά κτίρια λοιπόν έχουν καταστραφεί στη Δυτική Όχθη και τι βλέπουμε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ποινή για τις πράξεις αυτές. Κυριαρχεί πλήρης ατιμορρησία. Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά επεκτείνει και τους επικισμούς του σε παλαιστινιακά εδάφη. Τι κάνουμε εμείς για αυτή την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, για την κατάφορη κατεδάφιση των ευρωπαϊκών αυτών κτηρίων, των κτηρίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο περίφημος αυτός διαρθρωμένος διάλογος, κυρία Μογκερίνη, είναι μια φάρσα, φαρσοκομωδία τελικά, δεν οδηγεί πουθενά και καταδεικνύει τελικά ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την ουσία του προβλήματος. Δεν μπορεί να σταματήσει επικισμού στη Δυτική Όχθη. Έχει έρθει λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου για να σταματήσουμε την ανεκτικότητα αυτή που δείχνουμε απέναντι στους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ας ακολουθήσουμε την απόλυτη αλήθεια όσον αφορά τις καταστροφές των κτηρίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας ζητήσουμε αποζημιώσεις και σταματήσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω παροχή βοήθειας από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση και να στείλουμε μια διερευνητική αποστολή αυτή τη στιγμή στη Δική Όχθη για να δούμε πραγματικά πώ έχουν τα πράγματα εκεί πέρα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια αποτίμηση τη κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί η κυρία Νταμάτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε πραγματικά για την Παλαιστίνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους που είναι υπέρ και κατά του Ισραήλ, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποτίθεται ότι θα πρέπει να περασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά προτεραιότητα. Άρα θα πρέπει να περασπίζεται την τήρηση του διεθνούς δικαίου χωρίς καμία εξαίρεση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μιλάνε για κατάφορη παραβίωση του διεθνού δικαίου, μιλάνε για παράνομε πράξει. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και ανταυτού βλέπουμε ότι συνεχίζει το Ισραήλ να κατεδαφίζει όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν παραβιάζεται μόνο η σύμβαση της Γενέβης κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά τίθεται να αμφιβόλο και να κινδύνω και η ίδια η λύση των δύο κρατών. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να αποκαταστήσουμε την κατάσταση. Η Παλαιστίνη βρίσκεται σε πραγματική απόγνωση, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει μια μη κυβερνητική οργάνωση που φέρει το όνομα Breaking the Silence. Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση Ισραηλινή, αποτελείται, απαρτίζεται από απόμακους του Ισραηλινού στρατού, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν την επίτευξη τη Ειρηνή και συνεργάζονται με την Παλαιστινιακή κοινότητα. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί για ένα λεπτό συνάδελφος Πρέτσερ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, το όνειρό σας είπατε είναι η λύση των δύο κρατών και τι κάνει και τι, πώς συνεισέφερε προς αυτό το στόχο κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε με καθήκον επισήμανσης των προϊόντων από την Ιουδαία και τη Σαμάρια επίσης σε σχέση με τα κτίρια όσον αφορά τη ζώνη C, τη ζώνη Γ. Γνωρίζετε ότι για αυτή τη ζώνη εξακολουθεί να είναι όπως και κατά το παρελθόν υπεύθυνο το Ισραήλ για την ασφάλεια σε αυτή τη ζώνη και για την λύση σε σχέση με, με την λύση δύο κρατών θα πρόκειται για αυτοκτονία, αυτοχειρία σε σχέση με το Ισραήλ λόγω της του γεωγραφικού αναγλύφου αυτής της περιοχής και το γνωρίζετε και εφόσον αυτά τα κτίρια ε, στη ζώνη Γ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ισραηλινές μπουλντόζες θα τα κατεδαφίζουν και θα τα κατεδαφίζουν, κατεδαφίζουν νόμιμα και επειδή εδώ αφορά αυτό το θέμα την ασφάλεια του Ισραήλ και πρέπει αυτό να είναι προς το συμφέρον όλων μας η ασφάλεια του Ισραήλ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Πρέτσε. Για ένα λεπτό η συνάδελφος παρακαλώ. Σα Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο, πλήρως απαράδεκτο, απολύτως απαράδεκτο. Περιέγραψαν όλοι οι προλαλήσαντες της κατεδαφής. Και πώς αυτές εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του 2015. Σας ζητώ να μην συγκληθεί η διάσκεψη για τη σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ μέχρι να επιληθεί το ζήτημα, μέχρι να σταματήσουν αμέσως αυτές οι κατεδαφίσεις και να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση δράση για να σταματήσουν εκτοπισμοί, για να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις. Ακόμα και κτηρίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη συμβολή της, Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αρκούν τα λόγια, δεν αρκούν οι καταδίκες τα λόγια όταν παραβιάζεται το διεθνώς, διεθνές δίκαιο και με πολιτικές και με οικονομικές ε, συνέπειες. Ευχαριστώ. με συνάδελφε Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Σκρίπεκ. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σύγκρουση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη είναι μια τραγωδία η οποία συνεχίζεται εδώ και πολλέ δεκαετίε. Και τώρα συζητάμε του εκτοπισμού και τι κατεδαφίσει ε, ακόμα και κτηρίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ακούω όμω είναι ανησυχία για του Παλαιστίνιου. Αλλά στην σύγκρουση υπάρχουν δύο πλευρέ και όταν συζητούμε θα πρέπει να συζητούμε και για τι δύο πλευρέ. Αναρωτιέμαι γιατί οι 278 επιθέσει κατά Παλαιστινίων από Παλαιστίνιους μάλλον, κατά Ισραηλινών τους τελευταίους μήνες δεν αναφέρονται στα διεθνή μίδια. Γιατί όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τη Συμφωνία του 1995, ο τομέας ε, Γ παραμένει ε, υπό πλήρη στρατιωτική και διοικητική, ε, διοικητικό έλεγχο του Ισραήλ και θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνυπογράψει αυτήν την ε, συμφωνία. Και σας ρωτώ, είπατε εκπρόσωπε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσκάπτει τη συμφωνία χρηματοδοτώντας παράνομες κατασκευές στην περιοχή αυτή και δεν θεωρείτε ότι στέλνουμε το λάθος μήνυμα και προς τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Ευχαριστούμε συνάδελφε Σκρίπεκ. Για ένα λεπτό συνάδελφος Βάγκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, κυρία Μογκερίνη. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για τα πολύ καλά αυτά εισαγωγικά λόγια τα οποία μας είπατε για το ζήτημα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω παρά μόνο ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η συζήτηση αυτή γίνεται τόσο αργά σήμερα. Αυτό δείχνει πραγματικά την αδιαφορία και την άγνοια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το πολύ δύσκολο αυτό ζήτημα. Δεν θα αναφερθώ σε στατιστικά δεδομένα, αναφέραν πολλά ήδη προλαλήσαντες. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι όσοι καταστρέφουν παλαιστινιακά σπίτια προσπαθούν να δικαιολογήσουν την δράση τους αυτή η οποία βέβαια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση στα πλαίσια του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εμείς θα πρέπει να καταδικάσουμε αυτή τη μορφή τρομοκρατίας. Το να καταδαφίζει κανείς σπίτια σημαίνει ότι βάλει κατά της ίδιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτό ούτε για το Ισραήλ, ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για το σύνολο της περιοχής, ούτε για καμία χώρα τελικά του κόσμου. Το μόνο το οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι στους Παλαιστινίους. Ευχαριστούμε. Στη συνέχεια ο συνάδελφος λέει Αρίγκ. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, στο όνομα του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένουν με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στην κατάσταση που αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Όλε αυτέ τι κατεδαφίσει, καταρχά, μόνο και μόνο ο επικισμό είναι ένα φαινόμενο παράνομο. Δεν μπορούμε επίση να επιτρέψουμε ότι υπάρχουν χιλιάδε Παλαιστίνοι και παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα σπίτια του. Δεν μπορούμε επίση να επιτρέψουμε την καταστροφή των κτηρίων αυτών, των υποδομών, των οικονομικών που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια. Ακόμα και στα πλαίσια της Παλαιστινιακής κοινότητας αλλά και στα πλαίσια του ίδιου του Ισραηλινού στρατού ανησυχούμε πλέον όλο και περισσότερο για τη δράση την επίσημη του Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβληθούν κυρώσει Αυτή η συνεχής καταπάτηση της δημοκρατίας και του άρθρου 2 τη Συμφωνία σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ θα πρέπει να μα οδηγήσει στην αναστολή τη συμφωνία αυτή μέχρι το Ισραήλ να αρχίσει να σέβεται το διεθνέ δίκαιο. Νομίζω ότι θα πρέπει επιγόντω να περάσουμε σε δράσει. Ευχαριστούμε κύριε Λέια Ρίκα. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Ντυρόν. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπατή Πρόσωπε, τον Ιούλιο Είχα επισκεφθεί με άλλους συναδέλφους ένα χωριό στην Παλαιστίνη. Και σας δείχνω τι έχει απομείνει σήμερα από αυτό το χωριό. Ερήπια, μόνο ερήπια. Όλα τα άλλα κατεδαφίστηκαν. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περίπου 600 κτίρια, σπίτια, σχολεία έχουν κατεδαφιστεί από τις αρχές του έτους μεγάλο μέρος αυτών των κτηρίων είχαν χρηματοδοτηθεί η κατασκευή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προστατεύσει τον πληθυσμό των ε, ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή ΣΥ. Το Ισραήλ δεν είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν όλους τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τους αναγκάσει να το πράξουν, πρέπει να τους αναγκάσουμε να σταματήσουν οι καταδεύσεις φύσης και πρέπει να πληρώσει για τις παράνομες πράξεις του με αποζημιώσεις στο Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντυρό. Τώρα για ένα λεπτό συνάδελφος Παρνιό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι με τον Αλάν Μπενέρα, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, σε μια σημαντική γαλλική εφημερίδα είχαμε υπογράψει, υπογράψει ένα άρθρο στα πλαίσια του οποίου λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή ποτέ δεν βρισκόμασταν τόσο μακριά από μια ειρηνική λύση. Ποτέ η κατάσταση δεν ήταν τόσο απεγνωσμένη. Σπάνια βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη αδιαφορεί τελικά τόσο πολύ για την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτά τα 500 κτίρια, τα 500 σπίτια τα οποία έχουν ε, κατεδαφιστεί από το Ισραήλ. Πάρα πολλέ δομέ, υποδομέ που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση. Υπάρχουν πάρα πολλοί Παλαιστίνοι αλλά και Ισραηλινοί που θέλουν την ειρήνη μόνο και μόνο. Είχατε συμμετάσχει κι εσείς ε, τον Μάιο στην σύνοδο αυτή που έγινε στο Παρίσι προκειμένου να δοθεί νέα όθηση στην δενευτική διαδικασία, προκειμένου να διηγηθούμε σε μια λύση δύο κρατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσει η ρητορική μίσους, είναι σημαντικό να σταματήσουν οι επικισμοί. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η τροποποίηση των σχολικών εγχειριδίων. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να διηγηθούμε σε ειρηνική λύση. Ευχαριστούμε τώρα για ένα λεπτό. Γκέρικε, παρακαλώ. Αξιότιμη Επίτροπε, Πρόεδρε, πρέπει να επαναληφθούν αυτά. Πρόκειται για την χρήση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των Βεδουίνων και υπέρ των κατοίκων της περιοχής Γάμα και όλα αυτά χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όσον αφορά τις Ισραηλινές αρχές. Αυτό λοιπόν παράνομο. Αν υποθέταμε λοιπόν ότι είχε, είχε κατεδαφιστεί κάτι σε σχέση με την ε, ίδια τη Γερμανία και αυτό οδηγούσε σε φυλακίσεις. Ερώτηση η κυρία Μογκερίνη. Εδώ τι γίνεται σε σχέση με την πίεση που ασκείται έναντι του εταίρου μας ε, Ισραήλ. Εδώ λοιπόν ε, σε σχέση με την ε, αντίδραση του Ισραήλ θα εξακολουθήσουμε να δεχόμαστε ότι εδώ με χρήματα των φορολογουμένων μας θα ανεγείρονται πάντα κτίρια τα οποία θα είναι παράνομα και παρότι η, το Ισραήλ έχει υποστεί όλες τις επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, βρίσκεται εδώ χωρίς οποιαδήποτε ε, εξέταση μια καταδίκη του Ισραήλ. Είναι δυνατόν αυτό. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος Σιλικιώτης. Το Ισραήλ να συνεργαστεί για την εξέβρεση λύση συνεχίζει τους επικισμούς, τις εκτοπίσεις των πληθυσμό και καταστρέφει στοχευμένα ακόμα και τα παραπήγματα που στήθηκαν με χορηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοπεδώνουν κάθε κατάλημα στο οποίο στεγάζονται οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε απάνθρωπε συνθήκε. κάνουν του Παλαιστίνου πρόσφυγε ξανά στην ίδια του την πατρίδα. το ισραήλ με τι εγκληματικέ του ενέργειε αποδεικνύει πω στρέφεται ενάντια σε κάθε προσπάθεια τη Ένωση για στήριξη των παλαιστινίων και πώ αντιστατεύεται κάθε ειρηνευτική προσπάθεια. Α γίνει λοιπόν επιτέλου κατανοητό πως δεν αρκούν οι διακηρύξεις και εκφραστικές καταγγελίες καινού περιεχομένου. αν η ευρωπαϊκή ένωση σέβεται τις αρχές και τις διακηρύξεις της πρέπει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης μέχρι ότου το ισραήλ πάψει να παραβιάζει το άρθρο δύο στο οποίο αναφέρεται ξεκάθαρα η υποχρέωση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. είναι εξωφρονικό. τη στιγμή που γίνονται τόσε συζητήσει για αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση η ευρωπαϊκή ένωση να διαφορεί απέναντι στου παλαιστίνιου. Ευχαριστούμε κύριε Σιλικιώτη. Ακολουθεί για ένα λεπτό συνάδελφος Τέιλορ. Oh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε. Μογκερίνη, θα... οι αυξανόμενες καταδαφίσεις από το Ισραήλ στον τομέα Γ που πλήττουν σχολεία, εργοστάσια, σπίτια, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε από τις αναφορές των αποστολών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στην περιοχή. Τους πρώτους μήνες του 2016 έχουμε διαπιστώσει ότι ο αριθμός των καταδαφίσεων Παλαιστινιακών σπιτιών είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των καταδαφίσεων κατά το 2015. Επομένως αυτό είναι μια ευθεία επίθεση στην λύση των δύο κρατών είναι ξεκάθαρο ότι ο διαρθρωμένος διάλογος δεν δουλεύει. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Και ρωτώ, κυρία Μογκερίνη, θα προχωρήσετε με τη σύγκληση του Συμβουλίου ε, Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και την επίσκεψη του κυρίου Νετανιάχου όταν συνεχίζονται αυτές οι κατα, ε, κατεδαφίσεις. Μήπως επίσης θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε ποια ήταν η αξία η οικονομική αυτών των ε, κατεδαφισμένων κτηρίων. Ευχαριστούμε συνάδελφε Για ένα λεπτό ακολουθεί ο συνάδελφος Καν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Βλέπουμε αυτή τη στιγμή όλο και μεγαλύτερα κύματα κατεδαφίσεων στην περιοχή αυτή, καθώς επίσης και κατηναστικές εκτοπίσεις τόσο στη Δυτική Όγδη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας. Βλέπουμε ότι ε, οι αριθμοί έχουν ενταθεί πάρα πολύ ανησυχητικά τους τελευταίους μήνες και η πρακτική αυτή ουσιαστικά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά παρόλα αυτά το Ισραήλ συνεχίζει τη δράση του αυτή και ουσιαστικά στρέφεται κατά και τον ίδιο των Ευρωπαίων πολιτών, πολιτών που έχουν χρηματοδοτήσει τα έργα αυτά. Κατά αυτόν τον τρόπο τίθεται να αμφιβόλει η διαβιωσιμότητα τη λύση των δύο κρατών. Θα πρέπει το Ισραήλ να αρχίσει να τηρεί το διεθνέ δίκαιο, αν πραγματικά θέλει την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί, κυρία, είπατε εκπρόσωπε, θα μα ενημερώσετε πραγματικά για το ποσό των αποζημιώσεων και θα ζητήσετε τι αποζημιώσει αυτέ από το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Καν. Ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία συνάδελφο Σακοράφα παρακαλώ. Κυρία Μογκερίνη, οι εξελίξει στα κατεχόμενα επιβεβαιώνουν, θα έλεγα, την παταγώδη αποτυχία τη ευρωπαϊκή πολιτική στην περιοχή. Η εγκληματική πολιτική του Ισραήλ συνεχίζεται με του επικισμού και τι κατεδαφίσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη να μεγαλώνουν την απόγνωση και το αδιέξοδο του πληθυσμού. Μόνο φέτο έχει απαλωτριώσει 7.500 στρέμματα στη δυτική όχθη για επικισμό και η Ευρώπη παρακολουθεί σαν θεατή. Σα λέει αυθαρσό ο κύριο Νετανιάχου ότι καταστρέφει χρηματοδοτούμενε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπιστικέ δομέ, γιατί κατασκευάστηκαν, λέει, παράνομα και εσεί συμπεριφέρεστε σαν να μην σα νοιάζει. Και μα λέτε ότι είστε υπέρ τη λύση των δύο κρατών. Αλήθεια, πέστε μου, σε ποιο έδαφο θα δημιουργηθεί το Παλαιστινιακό κράτο. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, ότι σε λίγο δεν θα έχει απομείνει τίποτα. Ξεκινήσατε δομημένο διάλογο και βάλετε προθεσμία έξι μηνών. Έχει περάσει ένα μήνα από την λήξη τη προθεσμία και δεν πετύχατε τίποτα και αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να κάνει το ισραήλ για να προχωρήσετε σε κυρώσεις σε βάρος του και να ενεργοποιήσετε τις ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχετε υποχρέωση να υπερασπίζετε σύμφωνα με τις συνθήκες ευρωπαϊκής ένωσης και που από ό,τι φαίνεται τις έχετε σαν διακοσμητικές συμφωνίες σύντασης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία συνάδελφε Σακοράφα. Ακολουθεί για ένα λεπτό συνάδελφος κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπατή εκπρόσωπε, αν είχα την πείρα εγώ και με... ήμουν ο ίδιος αυτόπτης μάρτης, δεν θα το πίστευα επισκέφθηκα κάποιους ομολόγους κοινοβουλευτικούς στη Δυτική Όφθη όπου είχαμε συζητήσεις η απελπισία εκφραζόταν στις τοποθετήσεις τους. Απεπισία, μια και η κατάσταση των Παλαιστινίων επιδεινώθηκε με την πάροδο των ετών. Αλλά αυτό που με εξόργησε ήταν η καταστροφή δομών κοινοτήτων που είχαν χτιστεί ή τουλάχιστον είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βεδουίνοι με τους οποίους συζητήσαμε μας έδειξαν τα ερήπια των αντισκήνων τους που πραγματικά ε, οι τακτίσματά τους είχαν καταστραφεί. Θα ήθελα να ξέρω κυρία Επίτροπε πόσο, με ποιο στένος θα ζητήσετε να αποζημιωθούν σε σχέση με τις καταστροφές που προκάλεσαν να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι από το Ισραήλ. Ευχαριστούμε κύριε Φρόιντα. Για ένα λεπτό Χουαρίστια Μπάουνθ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι προφανές ότι οι εκτοπισμοί και οι κατεδαφισμοί συστηματικοί των ε, κτηρίων στην υποκατοχή η Περιορδανία είναι μέρος της πολιτικής του Ισραήλ. Προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν βομβαρδισμούς και καταστράφηκαν και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μηδενική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ε, ηχθείως σε σχέση με την ε, κατοχή της λωρίδας της Γάζας, την κατάσταση κατοχή στην οποία ε, περνά η λωρίδα της Γάζας από τους Ισραηλινούς. Δεν εξυπηρέτησε σε τίποτα αυτή η στάση και είπατε ότι δεν πρέπει εδώ λόγια να λέγονται, αλλά υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένων δράσεων. Πολύ καλά. Οι συνάδελφοι Άντερσον και Άουκεν και άλλοι είπαν ότι πρέπει να πάψει πια η ατιμορρησία του Ισραήλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Χουαρίστια Μπάουνθ. Για ένα λεπτό η κυρία Αρένα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ κύριε Μογκερίνη γιατί δεσμεύεστε για τη Μέση Ανατολή και καταβάλλετε πάρα πολλέ προσπάθειε για την επίλυση τη διένεξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Συμφωνώ απόλυτα με το στόχο σα. Να καταφέρουμε με κάθε δυνατό τρόπο να διευκολύνουμε την ειρηνευτική διαδικασία και να καταφέρουμε να καταλήξουμε στη λύση των δύο κρατών. Σήμερα είπατε ότι επικεντρωνόμαστε σε μία μόνο πτυχή της διένεξης αυτής. Δηλαδή, καταστροφή υποδομών έκτακτης ανάγκης, πρώτης ανάγκης που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παλαιστινιακό έδαφος. Μου κάνει εντύπωση οι ορισμένοι συνάδελφοι εδώ πέρα δεν βλέπουν την πραγματικότητα οι υποδομές αυτές δεν είναι παράνομες, οι επικισμοί είναι παράνομοι, οι επικισμοί θα πρέπει να σταματήσουν. Επομένως να λέμε ότι οι ανθρωπιστικές υποδομές που πληρώθηκαν από εμά είναι παράνομες, αυτό πραγματικά θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές. Αυτό το οποίο λοιπόν ζητάμε εμείς είναι να καταφέρουμε να ανακτήσουμε το διάλογο, να καταφέρουμε να επιβάλλουμε αν κρυθεί αναγκαίο κυρώσει και να καταφέρουμε να έχουμε και κάποιε αποζημιώσει αν το κρίνουμε αναγκαίο. Σας ευχαριστούμε κυρία συνάδελφε Αρένα. Ακολουθεί για ένα λεπτό η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Τον προηγούμενο μήνα είχα πάει στη Δυτική Όχθη, στη Δυτική Ιερουσαλήμ και είδα το τι συνέβαινε. Με ανησύχησε πάρα πολύ η κατάσταση εκεί όσον αφορά και την ίδια την διαδικασία ερήνευσης ε, για τη δημιουργία δύο κρατών που θεωρούν όλοι αναπόφευκτοι σε σχέση με κατεδαφίσεις ε, και εκτοπισμούς ε, και την ταπείνωση που συνεχίζεται με ασύνετο τρόπο, με βλακώδη τρόπο από το Ισραήλ Τίποτα καλύτερο για να προαθεί η ριζοσπαστικοποίηση των παιδιών της Παλαιστίνης στο μέλλον. Και σε σχέση με τους Βεδουίνους, ε, σε σχέση με την καταστροφή κτηρίων και κατεδάφιση τους ε, με χρήματα των Ευρωπαίων ε, φορολογουμένων δημιουργήθηκαν. Κυρία Μογκερίνη, θα έπρεπε να σταματήσουν αυτές οι δράσεις. Ζητήθηκαν ήδη αποζημιώσεις από το Ισραήλ για την καταστροφή δομών και κτηρίων που χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Πραγματικά εδώ ανησυχούμε για την ε, ανασφάλεια που δημιουργείται, για τη δική μας ασφάλεια και άλλο κόστος εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ειρήνευση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ είπατε εκπρόσωπε. Σήμερα παρακολουθήσαμε μία σουραλιστική συζήτηση. Αντί να μιλήσουμε για τους Ισραηλινούς εκείνους οι οποίοι δέχονται τόσες πολλές επιθέσεις ε, βίας, συζητήσαμε κάτι εντελώ διαφορετικό αντί να μιλήσουμε για το τσιμέντο αυτό το οποίο αποτελεί πολλές φορές αντικείμενο κλοπής για να χτιστούν αυτά τα τούνελ του τρόμου, μιλάμε για κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά Παλαιστινίων τα οποία πολλές φορές παίρνουν μαχαίρια στα χέρια τους και επιτίθενται στους ε, Ισραηλινούς. Μιλάμε για πραγματικά φαινόμενα αντισημιτισμού. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε φορά που τροφοδοτεί με τον ένα τον άλλο τρόπο τον αντισημιτισμό οδηγείται τελικά στην τρομοκρατία. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με κάτι σοβαρό. Όλα αυτά τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή οι ίδιοι Ισραηλινοί. Ένας μεγάλος αριθμός των οποίων δολοφονήθηκε μόνο και μόνο αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε συνάδελφε Ματουσέλο. Συνάδελφε, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σε λίγες ημέρες θα αποτίσουν το φόρο στα ε, θύματα του λογοκαυτώματος Ισραηλινή και θα γιορτάσουν ε, το τέλος του πολέμου των 7 ημερών. Επομένως είναι μια ε, κατάλληλη στιγμή για να αναρωτηθούν για την πολιτική τους. Αυτές τους τελευταίους μήνες έχουν κατεδαφιστεί σχολεία, νοσοκομεία, έχουν, οδηγήσει πολλούς Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τις αισθίες τους θα πρέπει να υποστηρίξουμε ε, εκείνους οι οποίοι μιλούν υπέρ της ειρήνης, υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και υφίστανται τις διώξεις ε, της Ισραηλινής κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι οι κατεδαφίσεις γίνονται σε στρατηγικά επιλεγμένους τομείς, τον ε1 κοντά στην Ιερουσαλήμ, για παράδειγμα. Αυτές οι ενέργειες του Ισραήλ ε, δημιουργούν κίνδυνο και υπονομεύουν τη δυνατότητα της επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος με τη λύση των δύο κρατών. Και αυτό για εμά θα πρέπει να είναι μια κόκκινη γραμμή. Θα πρέπει να απαιτήσουμε αποζημιώσει για τις καταστραμμένες υποδομές που χρηματοδότησε η Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Βόρτ. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ κύριε πρόεδρε Δεδομένη της καθημερινής και αυξανόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρατηρούμε στη δυτική όχθη είναι ανάγκη να δοθεί άμεσα λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα. φέτος μόνο ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει ολοσχερώς περίπου τετρακόσια οικίματα και άλλα κτίρια που κατασκευάστηκαν με κονδύλια της ευρωπαϊκής ένωσης στη δυτική όχθη ενώ πρόσφατα κατεδάφισε ένα σχολείο στην περιοχή γεγονός που σημαίνει ότι 23 παιδιά δεν θα πάνε πλέον σχολείο επιπλέον ο ε, ισραηλινός στρατός προχωρά στην κατάσχεση των εδαφών των παλαιστινίων και περιορίζει τις κινήσεις τους όσων ζουν στα κατεχόμενα εδάφη παράλληλα οι εκτοπισμοί πληθυσμού στην περιοχή είναι διαρκείς ενώ ο παλαιστινιακός πληθυσμός στη δυτική όχθη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νερού εξαιτίας της χρήσης του μεγαλύτερου ποσοστού αυτού του νερού από το ισραήλ και τους ισραηλινούς επίκους. είναι επομένω αναγκαίο να επιληθεί άμεσα το παλαιστινιακό ώστε να έχουμε βιώσιμη λύση και στη μέση ανατολή. η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια για την καταπολέμηση της φτώχειας στην περιοχή τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαρία. Ουρμπάν Κρέσπο παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η ευρωπαϊκή κοινωνία ζητά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να λογοδοτούν τα θεσμικά όργανα και να έχουν συγκεκριμένα προγράμματα δράσεων με στόχο να πάψει πια η κατοχή και να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση μακροπρόθεσμη σε σχέση με τον τερματισμό του Απατχάιτ που υφίστανται οι Παλαιστίνοι. Ζητούμε από την ύπατη εκπρόσωπο να απαιτήσει από την Ισραηλινή κυβέρνηση την πάψη των εκτοπισμών και την καταστροφή και τους κατεδαφισμούς ε, καθώς επίσης ε, και την επέκταση των οικισμών ε, των επικιστών Ισραηλινών στην Υπεριορδανία. Τέλος, ζητούμε σαφή τοποθέτηση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι αρχές του Ισραήλ καταστρέφουν δομές ανθρωπιστικού χαρακτήρα με χρήματα που οικοδομήθηκαν με χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Οι διαρκείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου ανθρώπου και της ε, διεθνούς νομοθεσίας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με την ένοχη σιγή ηχθείως των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Να επιβάλλετε κυρώσεις, να πάψει ατιμορρησία. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Ακολουθεί για ένα λεπτό συνάδελφος Μαραγκάλι παρακαλώ. Μικρό. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Yes. Μάλιστα, κυρία Μογκερίνη, εδώ και δύο χρόνια αναφέρθηκε ότι είπατε η προτεραιότητά σας ήταν η σύραξη Παλαιστινίων Ισραηλινών. Το είπατε αυτό ευθύ εξ αρχής. Τα αποτελέσματα είναι περισσότερο ε, εξόφθαλμα. Ακόμα μεγαλύτερη βία, ακόμα μεγαλύτερες παραβι... περισσότερες παραβιάσεις γελιοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κτίρια και οικήματα έχουν καταστραφεί και κατεδαφιστεί χωρίς προηγούμενο. Όχι μόνο τα σχολεία, γιατί παράνομα είναι τα όπλα και οι μπουλντόζες, όχι τα σχολεία, οι μπουλντόζες και τα όπλα που κατεδαφίζουν και καταστρέφουν. Εδώ υπάρχει χρεοκοπία, όχι δική σας προσωπική, αλλά χρεοκοπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ πήγα εκεί και είδα τι συνέβη με τους Βεδουίνους. Και εδώ πρέπει όταν αναφέρθηκε ότι η λύση δεν είναι να τακτοποιηθεί η κατάσταση των Βεδουίνων, αλλά να καταστραφούν τα οικήματά τους ε, όπου βρίσκονται σε υποέλεγχο των Παλαιστινίων. Σήμερα τηρούμε συγγύνη ηχθείως όσον αφορά την επέκταση των επικισμών των Ισραηλινών. Τι θα κάνουμε, θα τερματιστεί η ατιμορρησία του Απαρτχάντη ή όχι. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μαραγκάν. Στη συνέχεια ο συνάδελφος Μπούχνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ είπατε εκπρόσωπε που προσήλθατε εδώ και ακούσατε τις απόψεις σας. Εγώ πέρσι πήγα στην Παλαιστίνη και πρέπει να πω ότι ε, με έπληξε αυτό οδυνηρά όχι μόνο για την καταστροφή υποδομών με αυθαίρετο τρόπο από τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς όχι. Οι φυλακές στο ίδιο το Ισραήλ είναι υπερπλήρεις από παιδιά και εφήβους. Επαναλαμβάνω, αποκρατούμενους παιδιά και εφήβους. Όταν βρέθηκα εκεί ένας νέος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ ε, υποτίθεται ότι επειδή είχε ρίξει μια πέτρα σε ένα τεθωρακισμένο και προσπαθούσε να διαφύγει τον πυροβόλησαν. Αυτό είναι μια εκτέλεση εξοδικαστική. Ο, εκείνος που πυροβόλησε ο Ισραηλινός τον επεφήμισαν ως ήρωα οι Ισραηλινοί. Θέλω να πω ότι με ένα κράτος που κάνει τέτοια εγκλήματα δεν μπορούμε να έχουμε προνομιακές σχέσεις και συμφωνίες. Δεν μπορούμε να δίνουμε όπλα και οπλισμό σε αυτό το κράτος. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί. Αν λέμε ότι έχουμε κάποιες αξίες που θεωρούμε ότι είναι υπεράνω όλων. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούχνερ. Εδώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία CASDI και θα λάβει για να ολοκληρωθεί η συζήτηση τον λόγο η, συνάδελ, η κυρία είπατε εκπρόσωπος η κυρία Μογκερίνη, η κυρία Επίτροπος Μογκερίνη. Παρακαλώ. Uh, σας ευχαριστώ. Απ' τη μία θέλω να σας πω ότι θεωρώ τιμή μου. Πιστεύουν ορισμένοι ευρωβουλευτές ότι μέχρι σε 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου θα μπορούσα να είχα επιλύσει το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό πρόβλημα. Μακάρι να μπορούσα. Ποιο ξέρει, ίσω τα επόμενα 3,5 χρόνια να το λύσω. Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει πρόοδο. Όμως, θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε να έχουμε ε, εστιασμένη την πολιτική μας και να παραμένει συνεκτικό το μήνυμα που αποστέλουμε. Γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στην περιοχή Είμαστε ο σημαντικότερος δωρητής προς τους Παλαιστίνιους, είμαστε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος ε, για τους Ισραηλινούς, αλλά επίσης θα έλεγα και είμαστε και ο μόνος ε, φορέας, ε, ο, μόνος οργανισμός στο διεθνές επίπεδο που έχουμε μια συνεχτική πολιτική στο πρόβλημα αυτό, το οποίο, η οποία μάλιστα προέρχεται από την ιστορία της Ευρώπης. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι λυπούμε. Όταν ορισμένες φορές διαπιστώνω ότι και ακόμα και στο Κοινοβούλιο υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν τη μία πλευρά ή την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι οι αρχές μας που είναι διαπραγμάτευτες μας, ε, πρέπει να είναι αυτές που μας οδηγούν. Ωστόσο πρέπει να είναι ξεκάθαρος και ποιος είναι και ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι εκείνος του γεφυροποιού. Πρέπει δηλαδή να βοηθήσουμε εκείνους που ακόμα προσπαθούν στο εσωτερικό των κοινωνιών τους, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, ε, να υποστηρίξουν τη δημιουργία της λύσης και την ειρηνική συνύπαρξη ε, και των δύο ε, λαών αυτών. Ήταν κάτι δεδομένο αυτό την εποχή των συμφωνιών του Όσλο. Εγώ ανήκω στην γενναία εκείνων των πολιτικών που θεωρούσε την συμφωνία του Όσλο κάτι δεδομένο, κάτι σημαντικό. Σήμερα όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες φωνές και στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη που θεωρούν ότι η κατάσταση σημερινή δεν μπορεί να διαωνιστεί, δεν είναι φυσιολογική και χρειάζεται να συνεργαστούν Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι. Και πιστεύω λοιπόν ότι ακριβώς αυτούς θα πρέπει να βοηθήσουμε και να διευκολύνουμε. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ και να ευχαριστήσω ε, εκείνους που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία των ε, μελών των κοινοβουλίων υπέρ της ειρήνης και η οποία ε, έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι και Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους βουλευτές που προσπαθούν να ε, εξευρεθεί μια ε, ειρηνική λύση. Γιατί εμείς δεν το θεωρούμε πρόβλημα. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να είμαστε φίλοι και με τους Ισραηλινούς και με τους Παλαιστίνιους και δεν βλέπουμε καμία αντίφαση σε αυτό. Γιατί διατηρώντας φιλικές σχέσεις και με τους δυο μπορούμε να ασκούμε πιέσεις, να ενθαρρύνουμε ορισμένες φορές ε, πιο ξεκάθαρα ορισμένες φορές, πιο διπλωματικά ε, τις προσπάθειες για ε, την ειρήνευση στην περιοχή. Βεβαίω, όπως σωστά είπατε, θα πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη, να συνεχίσουν να εμπιστεύονται και οι δύο πλευρές την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της στην περιοχή. Θα ήθελα εγώ να σας αναφέρω κάτι το οποίο έγινε πρόσφατα και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο κύριος Νετανιάχου έδωσε εξαιρετικά ενθαρρυντικά μηνύματα και ακόμα και, και είπε ότι ακόμα και σε θέματα στα οποία δεν έχουμε συμφωνή ταύτιση απόψεων μπορούμε να συνεργαστούμε για να βρούμε κάποιον κοινό τόπο. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε, να χτίζουμε γέφυρες. Τούτου λεχθέντος όμως. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο ρόλος μας. Η πολιτική μας θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη και είναι απολύτως ξεκάθαρα διατυπωμένη και έναντι των Ισραηλινών και έναντι των Παλαιστινίων. Επίσης έχουμε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει πλήρης ενότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κανείς δεν θα καταφέρει να μας διχάσει ε, ούτε στο επίπεδο των κρατών μελών, ούτε στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων. Αυτό το έχω επαναλάβει πολλές φορές. Και ποια είναι αυτή η πολιτική μας. Η πολιτική μας λοιπόν είναι ξεκάθαρα εξή. Είμαστε εναντίον των επικισμών, είμαστε εναντίον της ρητορικής τους μίσους, είμαστε εναντίον της βίας. Επίσης, τα έργα αυτά τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη θεωρούμε ότι κατασκευάστηκαν για έναν ε, λόγο και μόνο έναν λόγο για το λόγο της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας ο οποίος, η οποία γίνεται με αμεροληψία και πλήρη ουδετερότητα και την ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να την παρέχουμε οπουδήποτε και οποτεδήποτε είναι απαραίτητη. Σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι και κάθετοι. Επίσης, θα το επαναλάβω, μιας και αναφέρθηκε από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, συνεργαζόμαστε ε, και με πολλά κράτη-μέλη για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα και στις δεχόμενα που εξετάζουμε η απέτηση αποζημιώσεων για τις ε, καταδαφίσεις. Αλλά τονίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι στο εσωτερικό μας, ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι ένα από τα ισχυρότερα μας ε, σημεία μέχρι στιγμής. Εμείς θέλουμε να επενδύσουμε στις δομές που μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζεται ο διάλογος και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τις αρχές του Ισραήλ. Πολλοί μου ζήτησαν να αξιολογήσω τους μηχανισμούς που δημιουργήσαμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής για αυτούς, γιατί παρά τα όποια προβλήματα χρειάζεται να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για να μπορούν να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, αυτές οι διαπραγματεύσεις με διαφάνεια και να συνεχίζουμε το διάλογο και με τους Ισραηλινούς και με τους Παλαιστινίους. Και κλείνω λέγοντας. ότι η πολιτική μας είναι η λύση των δύο κρατών. Αυτό ίσως μπορεί να μην το δούμε τον επόμενο 1,5 χρόνο. Δεν μπορώ να το υποσχεθώ. Αλλά αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το κουαρτέτο, το οποίο παρεμπιπτόντως να υπενθυμίσω ότι πριν από 1,5 χρόνο που ανέλαβα καθήκοντα δεν λειτουργούσε, ουσιαστικά, Συνεχίζουμε λοιπόν την συνεργασία με το Κοτέτο και στην έκθεση στην οποία προετοιμάζουμε θα αναφερθούμε εκτενώς στο θέμα. Επίσης συνεχίζουμε τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία, με τον ε, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με ε, τρίτες χώρες, ε, αραβικές χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις. Και προετοιμάζουμε και μια, ε, έναν κατάλογο συστάσεων, προτάσεων που η διεθνή κοινότητα θα μπορούσε να υποβάλει στα ε, εμπλεκόμενα μέρη. Βεβαίω δεν υπάρχει μια μαγική λύση που θα δημιουργήσει αύριο δύο κράτη και θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά ε, χαίρομαι για το γεγονό ότι η ειρηνευτική διαδικασία αναθερμάνθηκε και ξεκίνησε πάλι να συζητείται του τελευταίους μήνες. Είμαι πεπισμένη ότι συνεργαζόμενοι με τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε θετικές εξελίξεις, σε θετικά αποτελέσματα. Το ξέρω ότι κάποιος όταν το αναφέρει αυτό στη σημερινή συγκυρία μπορεί να ακούγεται ίσως υπερβολικά αισιόδοξο. Αλλά εάν δεν αναλαμβάνει κανείς το ρίσκο να αλλάξει την πραγματικότητα δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Γι' αυτό σας ζητώ να συνεργαστούμε, να υποστηρίξετε και εσείς από την πλευρά σας ε, και να διευκολύνετε τις προσπάθειες που γίνονται, γνωρίζοντας ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη έναντι και των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, κυρία Μογκυρίνη.